που είναι εδώ παρόν για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Και δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον κύριο Λαμασού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια είναι η πρώτη φάση της καινούργιας περίοδου για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη ή ότι διαπιστώνουμε ότι διότι ανάπτυξη σιγά σιγά μπορεί να ξαναρχίσει στην Ευρώπη, μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου, η ισοτιμία του ευρώ είναι χαμηλότερη και η Κεντρική Τράπεζα καθώς και η ΕΤΕ και το σχέδιο Juncker μας ενισχύουν σε αυτές μας τις εντυπώσεις. Θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη πρώτα χρησιμοποιώντας περισσότερα ποσά που να επενδύονται στην Ευρώπη από το εξωτερικό μέσω βέβαια μεγαλύτερης σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφαιρώντας τους φραγμούς που υπάρχουν ακόμη μεταξύ χωρών μελών για τις επενδύσεις. Αυτό είναι όλο το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης εξάλλου. Βασιστήκαμε καταρχήν μαζί με την Κομισιόν σε μία ανησυχητική διαπίστωση. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια που διατίθενται στον κόσμο αλλά όχι για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και πολύ λίγα από αυτά κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις εμποδίζονται γιατί έχουν υπερχρέωση και δεν μπορούν να υποφεληθούν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν συντηρητική πολιτική ή επενδύουν εκτός Ευρώπης και οι τράπεζες εξαρτώνται υπερβολικά συχνά ακόμη από τις κρατικές επιχορηγήσεις και βοήθειες. Όσοι λοιπόν θέλουν να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη δεν έχουν πάντοτε τον τρόπο να το κάνουν αυτόνομα και δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που σαν κάποιο επενδυτικό ταμείο όπως προτείνουμε που να τα διευκολύνει όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη της αγοράς και ένα νέο μέσον επένδυσης των υπαρχόντων ποσών όπως των εταιριών που δεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο καθώς και από τα ευρωπαϊκά ταμεία παρακινδυνευμένων κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια. Αυτού του είδους τα κεφάλαια θα έπρεπε να δεχτούν βέβαια να παγώσουν τις επενδύσεις τους κατά κάποιο χρόνο ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές ανα πάσα στιγμή να αφαιρέσουν, να επιστρέψουν τα κεφάλαιά τους αλλά με λιγότερα επιτόκια βέβαια. Ορισμένοι επενδυτές που, και εταιρείε που επενδύουν το κεφάλαιό τους κατά λιγότερο από 70% θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυστηρότερους κανόνες και μεγαλύτερη σταθερότητα ώστε να μπορούν με καθορισμένο χρονικό διάστημα να διοικούν ασκούνται να επενδύουν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης επιστροφής των κεφαλαίων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο ελαστικά ώστε να συμπεριλάβουμε και τα hedge funds και τα κεφάλαια ιδιωτών. Είναι δύσκολο βέβαια τα επενδυτικά ταμεία όπως ε, τα συνταξιοδοτικά και ορισμένα ε, κοινοτικές αρχές να πιστούν αλλά θα το προσπαθήσουμε. Θέλουμε να υπάρξει έτσι ένα ολόκληρη εργαλειοθήκη επενδυτική στην Ευρώπη που να αρχίσει να λειτουργεί μαζί με το σχέδιο Juncker για την αύξηση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Επίτροπος Βέσταγκερ. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαιρετίζουμε αυτή την θετική προσέγγιση για το ζήτημα που είναι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι μας έχει όλους πείσει ο κύριος Λαμασούρ, ο εισηγητής. Τον ευχαριστούμε θερμά, αλλά και την κυρία Κράτσα που δούλεψε κατά την προηγούμενη κοινωνική θητεία. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει την πρόθεση συμβασμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα όπως ε, ε, όσον αφορά αυτή την ποσόστοση των επενδύσεων γιατί έτσι ε, θέλουμε να δώσουμε τέτοια μορφή επενδύσει που να είναι ελκυστικές και για τους διαχειριστές και για τους επενδυτές. Και αυτά τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, τα ΕΜΕΚ, έχουν να κάνουν με κάποια στοιχεία ενεργητικού, με στοιχεία υποδομής, ε, μακροπρόθεσμα έργα και προγράμματα, μη συγμένε εταιρείε, εισηγμένε εταιρείε και μέχρι κεφαλαιοποίηση 500.000 αλλά και δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ούτω ώστε αυτοί οι διαχειριστές να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα σε πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ούτω ώστε όλα αυτά να διέπονται από ένα στεγανό νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό και είναι σημαντική η δουλειά μας ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη βοήθεια των χρηματοοικονομικών αγορών στην πραγματική οικονομία. Να, επομένως τώρα μια συγκεκριμένη έκφραση του τι κάνουμε για τις κεφαλαγορές, διότι σήμερα οι ιδιώτες επενδυτές ε, θέλουν να επενδύουν μακροπρόθεσμα και έχουν να αντιμετωπίσουν κατάτμιση των εσωτερικών αγορών ε, είτε σε συγκεκριμένη χώρα, κατάτμιση, είτε θέλουν να δράσουν διασυνοριακά. Οπότε βλέπουμε το ότι τώρα μπορούμε να έχουμε περισσότερες θετικές ε, συνέπειες των επενδύσεων και για την απασχόληση και για την οικονομία. Οπότε τώρα λύνουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε τώρα κανόνες ομοιόμορφους και έτσι όλοι οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν για τις ΜΜΕ, για κάποια μακροπρόθεσμα έργα και προγράμματα και έτσι έχουμε το πρώτο βήμα για μια άλλη ένωση κεφάλαια αγοράς. Ούτως ώστε τώρα να έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων. Και γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αυτό τη σήμερα ημέρα είναι ακόμα πιο σημαντικό, όπως το είπε ο κύριος Λαμασούρ. Τα πράγματα τώρα είναι κάπως πεσμένα, με την ισοτιμία του ευρώ, την κρίση κλπ. Όμως χρειάζονται οι επενδύσεις. Και 1,5-3 είπαμε θα έχουν γίνει επενδύσεις μέχρι το 2020. Ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν τα, αυτά τα έργα υποδομής τα οποία τα χρειάζονται τόσο πολύ. Οπότε αυτά τα ΕΜΕΚ εδώ θα διαμετούν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της οικονομίας, εκεί που θα έχουμε δέσμευση μακροπρόθεσμη του κεφαλαίου. Και εμείς επομένως έχουμε δεσμευθεί σε αυτό τον τομέα και αυτό βέβαια δεν βγάζει τη τράπεζα από το παιχνίδι γιατί οι τράπεζες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των έργων σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε και γι' αυτό τα ΕΜΕΚ θα παίξουν συμπληρωματικό ρόλο σε αυτή την δραστηριότητα. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ανέκαθεν συμφωνούσαν ότι οι ΜΜΕ έχουν μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και το να χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτά τα στοιχεία ενεργητικού για τις επενδύσεις είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως θα πρέπει να σας επενέσω, γιατί εδώ και υλικά στοιχεία περιουσιακά, αλλά και στοιχεία πνευματικής διοκτησίας τα έχετε συμπεριλάβει. Πολύ σημαντικό όλα αυτά για τις οικονομίες μας, οπότε χρειάζεται τώρα αυτή η χρηματοδότηση ακριβώς, όπως και τα έργα υποδομής. Οπότε τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το πώς θα ελκύσουμε και θεσμικού επενδυτέ και μεμονωμένους επενδυτέ, και στη εξωτικά ταμεία. Όλοι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ΕΜΕΚ γιατί αυτό πάντοτε ήταν ε, κλειδί στις δικές μας προτάσεις. Το ότι εσεί. θέλετε να υπάρχει προσημότητα και από μεμονωμένους επενδυτέ, είναι πολύ σημαντικό ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Επίσης, μπράβο σας που θέλετε να έχουμε αυτές τις ιδιαίτερες ρήτρες διαφύλαξης, ώστε να επιτρέψουμε στου επενδυτέ κάτω του μισού εκατομμυρίου σαν περιουσία για να μην ε, βάλουν παραπάνω από 10% των αποταμιεύσεών τους σε τέτοια ΕΜΕΚ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και για την προσοχή σας. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να λαμβάνετε υπόψη την ανάγκη σεβασμού του χρόνου σας. Γιατί όπως ξέρετε πρέπει η ψηφοφορία να αρχίσει οπωσδήποτε στις 30 επειδή θα έχουμε και την επίσημη συνεδρίαση με τον ε, βασιλέα της Ιορδανίας στις 12. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Χιμπνερ. Ευχαριστώ. Για χρόνια τώρα μειώνονται και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Η προσπάθεια λοιπόν να υπάρξει χρηματοδότηση ανάπτυξη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κάνουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να προωθηθεί το σχέδιο Juncker ώστε να τον ταχύτερα από ιδέα σε πραγματικότητα. Και γι' αυτό όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμεθα για να δημιουργηθεί αυτό το LTIF ω θέμα ε, επίγουσα προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε μια κεφαλαϊκή αγορά με τρόπο που να αξιοποιεί τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να επιτύχει μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων ανάπτυξη. Αλλά φυσικά για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε το σωστό πλαίσιο. Για χρόνια προσπαθούμε να επιτύχουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τώρα πρέπει μέσω αυτής της σταθερότητας να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Αλλά αυτή η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα. Και γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν τα υπάρχοντα ακόμη, τα εναπομείνοντα ε, εμπόδια στην χρηματοπιστωτική ενιαία αγορά και όλες οι ατέλειες στην κεφαλή αγορά. Και το μήνυμα νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές. Πρέπει να γίνει μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από όλες τις πλευρές, τόσο στο ρυθμιστικό, όσο και στο μεσολαβητικό, όσο και στο επίπεδο των χρηστών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κόφοντ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης της ομάδας μου θα ήθελα να διασφαλίσω τη δημιουργία ενός ταμείου που να ωφελεί την πραγματική οικονομία και νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται έτσι. Η μακρά οικονομική κρίση και η έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη επενδύσεων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βελτίωση της οικονομίας και γι' αυτό το σχέδιο Juncker, το επενδυτικό σχέδιο Juncker και η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου θα βοηθούσε πολύ στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικό εργαλείο για την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη. Θα ήταν χρήσιμο παραδείγματος χάρη για ασφαλιστικές εταιρείες, για συνταξιοδοτικά ταμεία που χρειάζονται έναν μηχανισμό συνδυασμένου, συνδυασμού των επενδύσεών τους με στόχο να χρηματοδοτηθεί έτσι μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη που είναι κάτι ουσιώδες διότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να είναι και οικονομικά σταθερή αλλά και αναπτυσσόμενη και ελπίζουμε ότι αυτό το ΕΛΤΙΦ θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς για αυτό το στόχο. Πάνω απ' όλα όμως ελπίζω ότι το Ταμείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση βιώσιμης και οικολογικής ανάπτυξης που θα έχει και θετικές επιπτώσεις και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά για την Ευρώπη στο σύνολό της. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με επενδύσεις στην πράσινη και βιώσιμη οικονομία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πράσινη ανάπτυξη για να μην περάσουμε τα οικολογικά μας προβλήματα και στις επόμενες γενιές. Επενδύσεις και για τους μελλοντικούς Ευρωπαίους λοιπόν Καλούμε λοιπόν και τους ιδιώτες και τους μη ιδιώτες επενδυτές να κάνουν χρήση αυτού του εργαλείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Όζοκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η Κομισιόν έχει δίκιο για το χρηματικό ότι προσπαθεί δηλαδή να προσελκύσει κεφάλαια για να επενδυθούν στην Ευρώπη όπου και να διαβιούν. Αυτά τα κεφάλαια, ιδεοδός, θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αλλά και για την έρευνα. Αυτά τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες επενδυτές όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία για να μπορέσουν έτσι να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους και μέσα και έξω από την Ένωση. Το έγγραφό μας δίνει και περιθώριο ελιγμών στους επενδυτές λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού επίπεδου επενδύσεων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο κύριος Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ καθώς και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τελικά καταλήξαμε νομίζω σε έναν ε, σωστό συμβιβασμό γιατί η Ένωση της Κεφαλαιαγοράς για την οποία μιλάμε και θα μιλάμε τις επόμενες εβδομάδες είναι θέμα ποικιλομορφίας, σεβασμού της ποικιλομορφίας γιατί οι επενδυτές πρέπει να έχουν επιλογή για το πού θα επενδύσουν ιδίω οι θεσμικοί επενδυτές θα έχουν πια ένα ταμείο που να τους επιτρέπει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όχι μόνο σε έργα υποδομών, αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μετόχους τους. Θα έχουν δηλαδή την ποικιλομορφία που χρειάζονται. Επίσης είναι ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές για την, να βρουν νέο, νέα είδη επενδύσεων. Βέβαια δεν τελειώνουν όλα έτσι. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά και οι τράπεζες, ακόμα και μερικοί ιδιώτες μεμονωμένοι θα πρέπει να συνεχίσουν να χορηγούν κεφάλαια για επενδύσεις. Θα πρέπει το ταμείο αυτό βέβαια να μπορεί να τους επιτρέψει να επενδύουν και να διασφαλίσει ότι η όλη ένωση της κεφαλαιαγοράς θα λειτουργήσει βιώσιμα. Ότι θα υπάρχει ισοτιμία και για τη φορολόγηση και όπως είπε και ο Επίτροπος Χίλ, όλα αυτά ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη όπως πρέπει, ώστε το Ταμείο αυτό μακροπρόθεσμων επενδύσεων να αποδειχτεί βιώσιμο και μακροπρόθεσμα και να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη μεγαλύτερης ποικιλομορφίας και στην αγορά κεφαλαίων μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ουρβάν Κρέσπο παρακαλώ, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο επενδύσεων που υπεβάλλει η Κομισιόν λέει ότι θα επιτύχει ε, θαύματα ανάλογα του Ιησού. Και λέει δηλαδή ότι τα 21 δισεκατομμύρια θα μας οδηγήσουν σε 315 δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων. Και ένα από τα προϊόντα κλειδιά είναι αυτό το ταμείο ΕΛΤΙΦ, στο οποίο θα μπορούν, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιούν και οι θεσμικοί και οι ιδιωτικοί επενδυτές. Όμως, οι ρυθμίσεις που μας παρουσιάζουν δεν περιέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις που να προστατεύουν τον τελικό στόχο του επενδυτή υπάρχουν πολλές πόρτες ανοιχτές που θα επιτρέψουν στα κεφάλαια υψηλού κινδύνου και στα κεφάλαια γήπες να επενδύσουν. Θέλουμε εμείς να έχουμε στόχο να βοηθήσουμε το λαό. Αυτή η μακροοικονομική πολιτική έχει επιτύχει. Στη χώρα μου έχουμε τις θλιβερές επενδύσεις που λέγονται preferentes, δηλαδή προτιμησιακές επενδύσεις. Αλλά τα προϊόντα αυτά τελικά δεν ήταν διαφανή και οδήγησαν στην καταστροφή δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Συνάδελφοι, αυτό το λανθασμένο ευρωπαϊκό New Deal που αποκαλείται σχέδιο Juncker είναι αυταπάτη. Δεν θα αναζωογονήσει την ανανεμική μας οικονομία. Αυτή είναι ο φιλελεύθερη πολιτική. Τα προϊόντα αυτά, ELTIF, πώς είναι δυνατόν σε τρία χρόνια να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι αξιόπιστο αυτό δεν είναι δυνατόν ε, τα θεσμικά μας όργανα να χρηματοδοτούν αυτήν την οικονομία του καζίνου, αυτές τις φούσκες που, παίζει, που παίζουν με, τα, ε, με τις αποταμιεύσεις των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λαμπέρ, ε, 3,5 λεπτά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, η Ευρώπη είναι πλούσια ήπειρος όχι μόνο μέσω ιστορίας και πολυμορφίας αλλά και οικονομικά. Αλλά παρόλα αυτά η Ευρώπη δεν καταφέρνει να κάνει επενδύσεις. Δεν καταφέρνει να ε, αξιοποιήσει τις προοπτικές του μέλλοντός της. Όμως η Ήπειρός μας έχει ανάγκη από επενδύσεις. Δηλαδή να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση με το σωστό και υπομονητικό τρόπο. Για παράδειγμα, να χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή μετάβαση. Μιλάμε για την Ενεργειακή Ένωση που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μα. Πρέπει να επενδύσουμε στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την καινοτομία. Αυτέ είναι οι προποθέσει ανταγωνιστικότητά μα. Να επανακτήσουμε του φυσικού μα ε, πόρου και να επαναφέρουμε την κοινωνική συνοχή μα. Και σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Αλλά δεν γίνονται αυτέ οι επενδύσει. Και γιατί? Γιατί εδώ και 20 χρόνια το δόγμα που κυριαρχεί απόλυτα είναι η δικτατορία της μεγιστοποίησης του βραχυπρόθεσμου κέρδους. 20 χρόνια χρηματοπιστωτικής απορρίθμισης και τα πάντα μετριούνται με το χρήμα και τα πάντα μετρούνται με το πόσο θα κερδίσει ο επενδυτής. Και ποιοι είναι οι επενδυτές, τα ταμεία, οι, οι ιδιώτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, οι οποίοι επενδύουν σε διάφορες εταιρείες για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Πώς να αποκληθούν ε, επενδυτές όταν και οι πιο συντηρητικοί σου λένε ότι δεν θέλουμε να κρατήσουμε καμία μετοχή άνω της πενταετίας. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν. Το κείμενο αυτό κύριε Λαμασούρ είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά ένα τόσο μικρό βήμα, απόλυτα μικρό βήμα. Θέλουμε να προσελκύσουμε τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αλλά με εκπλήσει το ότι το Συμβούλιο, όπως υπογράμμισε και η κυρία Βεστάγκερ, αρνήθηκε αυτήν την ε, ποσόστοση επενδύσεων στην Ευρώπη. Είχαν πει ότι για να είναι κάποιο ταμείο, ε, ταμείο τύπου ΕΛΤΙΦ, 60% των επενδύσεών του έπρεπε να είναι στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο είπε ότι αυτή είναι κόκκινη γραμμή, δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Μα τι θέλει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει να ευνοήσει τους επενδυτές ή τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Αρνούμενοι την ευρωπαϊκή ποσόστοση, οι κύριοι και οι κυρίες του Συμβουλίου απέδειξαν από ποια μεριά είναι. Αν θέλουμε πραγματικά αναζωογόνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη θα χρειαστούν όμως και άλλα μέτρα. Πρώτη, πρώτο μέτρο θα είναι, πρέπει να είναι οι τράπεζες για τους ε, καταθέτες να είναι διαφορετικές από τις επενδυτικές τράπεζες. Εάν υποχρεώσετε να γίνονται επενδύσεις στην πραγματική οικονομία κλείνοντας δυνατότητες τύπου καζίνο, τότε θα βοηθήσετε την αζωγόνηση. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα λεγόμενα επενδυτικά προϊόντα που θέλουν να στύψουν ω λεμονόκουπα τον πλανήτη και του ανθρώπου του για την μεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου κέρδου. Πρέπει επιτέλου να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων. Και να σα δώσω δύο στοιχεία. 13 δι υπόσχεται δημόσιες επενδύσεις το σχέδιο Juncker 13 δις. Είναι το 1% της φοραπάτης και φοραπαλλαγής στην Ευρώπη. Αν ήμασταν σοβαροί στην καταπολέμηση της φοραπάτης και φοραπαλλαγής θα είχαμε χίλια δις, ένα τρεις δηλαδή, που θα έμπαιναν στο δημόσιο κορβανά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μπλε κάρτα, κύριε Λαμπέρ, από τον κύριο Έθερη. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Ευχαριστώ, μα πάντα ε, με καλή θέληση δέχεστε τις μπλε κάρτες. Μας είπατε πολλά, λέει ο κύριος Έθεριτς, για δημόσιες επενδύσεις και κρατικά κεφάλαια. Δεν θα συμφωνούσατε Ξέρω ότι αντιμετωπίζετε τα, το ιδιωτικό κέρδος αρνητικά, αλλά αν δεν υπάρχει ιδιωτική δημιουργία πλούτου και ιδιωτικό κέρδος, τα ταμεία αυτά που θέλετε να αξιοποιήσουν τις δημόσιες επενδύσεις δεν θα υπήρχαν. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ιδιωτική δημιουργία πλούτου επίσης μέσω για παράδειγμα μείωση της φορολογίας όπου γίνεται. Λαμπέα. Ε, ναι, έχουμε τη συνήθεια να συζητάμε. Ναι, συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι 100% της οικονομίας πρέπει να είναι δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις. αυτό ήταν το τελευταίο που είπα. Αλλά επίσης είπα ότι πρέπει οι τράπεζες να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Γιατί, Γιατί θέλουμε οι εξοικονομήσεις ε, των μεμονωμένων καταθετών να επενδύονται στην πραγματική οικονομία. Ναι, θέλουμε ιδιωτικέ επενδύσει, αλλά τι έχω δει στα 22 χρόνια που εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ότι ο χρονικό ορίζοντα των ιδιωτικών επενδυτών Μικραίνει συνεχώς. Συνέχεια. Ούτε καν ένα τρίμηνο, μια εβδομάδα, ένα χιλιοστό δευτερολέπτο. Μα δεν είναι επένδυση αυτή. Ναι, θέλω ιδιωτική επένδυση. Και βεβαίω είναι νόμιμα τα ιδιωτικά κέρδη, αλλά πρέπει να δημιουργούν αξία για την κοινωνία. Στίβεν Γούλφ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τζότζε Φάντισον, ήταν ένα πύρη που έλεγε ότι τον φοβάται κανεί τον θάνατο, πολλέ φορέ αυτό ε, σκοτώνει. Ε, και έτσι γίνεται. Και πολλοί προσπαθούν να σώσουν το τομάρι του και τελικά αυτό καταστρέφονται. Να βλέπω τι γίνεται και εδώ πέρα ο φόβος για την Ελλάδα τελικά έχει ρίξει το ευρώ, ο φόβος για την χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης έχει σκοτώσει την οικονομία και άρα βλέπουμε ότι τελικά απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά ήταν μια κακή ιδέα και τελικά έφαγε τα ψωμιά της. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι τώρα κάτι το οποίο τελικά θα οδηγήσει στην καταστροφή. Να, ακριβώ αυτή η στρατηγική για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, τα ΕΜΕΚ. φαίνεται, πιστεύει το Κοινοβούλιο ότι μπορούν κάποιοι τραπεζίτες να τονώσουν την οικονομία και γι' αυτό και η Κεντρική Τράπεζα έφερε αυτή την ποσοτική χαλάρωση που πρόκειται να εξασφαλίσει το ότι θα βάζουμε πιο βαθιά το για τη στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Τι γίνεται, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα έπρεπε τα κράτη να φτιάχνουν τηλέφωνα, δεν θα έπρεπε να φτιάχνουν ε, κομπιούτερ ή οι Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο πρετανεύει άποψη ότι οι βουλευτές και οι επίτροπες μπορούν να φτιάξουν τέτοια επενδυτικά ταμεία και μπορούν να γίνουν επενδυτές. Να, τι προϊόν τώρα προτείνεται. Μα σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι στον κόσμο των επενδύσεων και έχουν αποτύχει. Και εσεί, κατά μείζον λόγο θα αποτύχετε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Και τώρα δίνει το λόγο στον κύριο Μπρίουα για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων έχει, είναι μια καλή ιδέα φαινομενικά. Παρόλα αυτά, το κατά πόσον χρειάζεται ένα τέτοιο ταμείο ενωσιακά δεν έχει αποδειχτεί. Μιλάμε για τραπεζική ένωση και η συμπληρωματική έκθεση λέει ότι αυτό το ΕΛΤΙΦ είναι η πρώτη φάση για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων που να κατευθύνονται προς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αλλά σε ποια βάση θα γίνει η σύγκληση πανευρωπαϊκά. Γνωρίζετε ότι διαφέρουν οι νομοθεσίες μας για τις χρηματαγορές. Έπειτα, βάζοντας το ταμείο αυτό υπό τον έλεγχο της Κομισιόν, κάνετε ακόμη ένα λάθος και κοροϊδεύεται τα κράτη-μέλη και την κυριαρχία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νίτερ Μάιερ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κυρίες και κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι νομίζω ότι ένα από τα καθήκοντά μας είναι να βελτιώσουμε, να δώσουμε λιγότερο κατακαιρματισμό στην ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν όντως σε επενδύσεις που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Επομένως το ΕΛΤΙΦ αυτό είναι καλή πρωτοβουλία και το σχέδιο Βιούνκερ γιατί θα αλλάξει τελικά την συνολική εικόνα και θα καταλήξει σε πραγματική ανάπτυξη. Όμως οι χρηματικές διευθετήσεις δεν είναι το μόνο εργαλείο που χρειαζόμαστε. Καταρχήν Υπάρχει το θέμα των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται σε ορισμένα κράτη για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε ένα βιώσιμο δρόμο. Αν δεν έχουν μπει σε αυτόν τον βιώσιμο δρόμο δεν μπορούν να γίνουν και πολλά για επενδύσεις ή θα αποτύχουν αυτές. Δεύτερον, η έλλειψη σταθερότητας των ρυθμίσεων και των νομικών συστημάτων μεταξύ χωρών μελών που υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και αυτό εμποδίζει τους επενδυτές και τέλος ότι η ενιαία αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί μια ενιαία αγορά είναι κάτι το ουσιώδες για να υπάρξουν ρεαλιστικά τέτοια σχέδια. Το η πρώτη δοκιμή θα ήταν βέβαια η βελτίωση του ρυθμιστικού συστήματος αλλά Δυστυχώς η φραγμή είναι ακόμη πολύ. Ελπίζω να λυθούν όλα το ίδιο αποτελεσματικά όσο το εύχεται ο κύριος Λαμασούρ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Περβάν Μπερές για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε. Μιλάμε εδώ για μια έκθεση που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί πολύ νωρίτερα. Όταν το 2007 ξέσπασε η κρίση πανευρωπαϊκά, όλοι είδαν ότι επρόκειτο για κερδοσκοπία και για έλλειψη χρημάτων στην Ευρώπη. Χρειάστηκε όλος αυτός ο χρόνος για να σταθεροποιήσουμε τις χρηματαγορές και να σώσουμε τις τράπεζες. Αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε κάποια μακροπρόθεσμη επένδυση στην Ευρώπη για να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει δημογραφική, κλιματολογική κλπ. Καλό το νέο λοιπόν. Ίσως αύριο το ε, ταμείο αυτό, το ΕΛΤΙΦ, να γίνει κάποιο νέο μνημείο της Ευρώπης που θα αποδείξει ότι μπορεί, είναι ικανή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των επενδύσεων, της έλλειψης επενδύσεων. Επενδύσεων βέβαια όχι κερδοσκοπικών και εκτός φορολογικών παραδείσων με σεβασμό δε των κανόνων του ΩΣΑ. Αυτό θα είναι η δοκιμή και θα δείξει αν όντως θα καταλήξει και σε περισσότερη απασχόληση, αν υπάρξουν πράγματι στρατηγικές επενδύσεις όπου να μπορούν να συμμετάσχουν και οι ιδιώτες. Επίσης πρέπει να πάρουμε μαθήματα. Ο τριμερής διάλογος για το θέμα κατέληξε την ημέρα που ανακοινώθηκε η έναρξη του σχεδίου Juncker και αυτό είναι σημαδιακό. Πρέπει επιτέλους να υπάρξουν τέτοιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ελπίζω όταν θα εξετάσουμε και το σχέδιο του Επιτρόπου Χίλ για την Ευρωπαϊκή Κεφαλαία Αγορά να τα εξετάσουμε όλα αυτά και να πρόκειται πράγματι για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ευχαριστούμε. Φων Στόρκ. Ένα λεπτό. Συνάδελφοι, το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο μας λείπει στην Ευρώπη. Το είπε και ο κύριος Γιούνκερ. Λέει υπάρχει τράπεζα επενδύσεων. Αυτό το νέο ΕΛΤΙΦ προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Να δούμε πίσω στο παρελθόν. Όταν πήγαινε καλά το ευρώ γινόντουσαν και επενδύσεις. Ξέρουμε όμως ότι αυτό ήταν ε, αυταπάτη. Η προβλέψιμη κρίση του ευρώ και το γεγονός ότι το μέλλον του είναι τόσο αβέβαιο δημιούργησαν μεγάλη αβεβαιότητα για τους επενδυτές οι επενδυτέ εξαρτώνται από τις αποφάσεις των πολιτικών οπότε δεν ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις λόγω αυτού ακριβώς του πολιτικού κλίματος. Το ΕΛΤΙΦ δεν θα καλύψει αυτό το κενό επενδύσεων δεν καταργεί την αβεβαιότητα που είναι ο πραγματικό λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί το ευρώ και οι προσπάθειες ε, ε, διάσωση του ευρώ δυσχεραίνουν την κατάσταση. Δεν χρειαζόμαστε κανένα νέο ταμείο. Πρέπει να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Το ευρώ πνίγει την Ευρώπη. Μόνο αν το καταλάβουμε αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Νικολάη Νορίγκα. Μισή Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα. Εάν τα συζητούσαμε αυτά πριν από 10 χρόνια, τότε θα συζητούσαμε για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα και για την βιωσιμότητα και τελικά τα συζητάμε σήμερα όμως θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση όσων συζητούμε το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσει έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια θα έχει πολύ δουλειά μπροστά της ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, την ΕΣΜΑ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που διαθεσεί της. Επίσης, έτσι, με πόρους δηλαδή, και βρικοδότης θα μπορέσει το ΕΛΤΙΦ, να λειτουργήσει καλά. Υπάρχουν εδώ πολλέ δυνατότητε τόσο να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Με αυτόν τον κανονισμό προβλέπεται ένα επενδυτή να μπορεί να μπλοκάρει την μακροπρόθεσμη επένδυσή του και να μπορεί να αποεπενδύσει νωρίτερα. Προσοχή όμως να μην έχουμε κάποια στρέβλωση του συστήματος και τελικά να μπορούν οι επενδυτές να μπορούν να διαλέξουν πού θα επενδύσουν και έτσι να κερδοσκοπήσουν. Δεν φαίνεται το αποτελεσματικό το ταμείο. Ενάμιση λεπτό κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε ένα ζωτικό θέμα των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό μεν, αλλά δεν συζητήσαμε την καρδιά του προβλήματος συνεχίζουμε να το αποφεύγουμε. Πρώτον, η κεφαλαιαγορά, η ένωση κεφαλαιαγοράς θα παίξει σημαντικό ρόλο άραγε για να υπάρξει χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την οικονομία του καζίνου τέτοιο πρότυπο θέλουμε να ακολουθήσουμε ή αντίθετα θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και το δόγμα να δημιουργήσουμε νέα μέσα επένδυσης. Αν δεν υπάρχουν νέα επενδυτικά πρότυπα δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι το δόγμα λέει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ερωτώ λοιπόν, αναρωτιέμαι, η παραδοσιακή σχέση τραπεζών και οικονομίας τι θα γίνει. Γιατί δημιουργούμε όλο και περισσότερα μέσα που να θέτουν την οικονομία σε κίνδυνο. Δεν λύνουμε έτσι το πραγματικό πρόβλημα. Τίποτα δεν κάνουμε για το πραγματικό πρόβλημα, τη ζήτηση. Πρέπει να προωθήσουμε την ζήτηση και να απαλλαγούμε από τη λιτότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστούμε ο κύριος Τζάνι Μάρκο. Αυτό θα έπρεπε να είναι ευκαιρία του να στείλουμε ένα μήνυμα ισχυρό για την ε, πραγματική οικονομία. Όμως τώρα ρισκάρουμε ακόμα ε, μια πτώχευση, μια αποτυχία, γιατί βλέπουμε ότι τώρα θα ωφεληθούν οι πολυεθνικές και οι κερδοσκόποι και για άλλη μια φορά ξεχνούμε τις ΜΜΕ και τους ε, επενδυτές και, συγγνώμη, και τους αποταμιευτές αυτό θα γίνει με την αγορά, γιατί η ταυτότητα της Ευρώπης είναι οι αποταμιευτές. Την Ευρώπη σιγά σιγά την ξεχνάμε και όλες οι προτάσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τονώσει την παραδοσιακή αποταμίευση. Έχουμε ξεχάσει το κοινωνικό πρόσωπό μας, οπότε τώρα οδηγούμαστε ε, σε, στρεφόμαστε μόνο στην κεφάλαια αγορά, εκεί που βασιλεύουν οι κερδοσκόποι. Τι γίνεται με τον παραγωγικό ιστό. Βλέπουμε ποια είναι η πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα. Βασιλεύουν οι κρυπτοκάρτε των Βρυξελών και έχουμε τώρα απομίμηση του αμερικανικού μοντέλου της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε εγκαταλείψει τις ΜΜΕ στην τύχη τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα. ο κύριος Γιώργος Κίρτσος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που συζητάμε είναι ιδιαίτερα θετική και συμπληρώνει ένα αναπτυξιακό πάζελ ε, το οποίο έχει φυσικά μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, λύνουμε συγκεκριμένα προβλήματα όπως είναι η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου αλλάζει η εικόνα και βελτιώνεται η προοπτική. για παράδειγμα έχουμε τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την εξυγίανσή του έχουμε τη σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού και των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου ιδιαίτερα των λεγόμενων χωρών της ε, περιφέρειας αν και δεν δέχομαι ακριβώς αυτή τη διατύπωση αλλά εν πάση περιπτώσει η πτώση του κόστους δανεισμού για παράδειγμα της ιρλανδίας και της πορτογαλίας κάνει πιο διαχειρίσιμο το χρέος απελευθερώνει πόρους για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. επίσης έχουμε υποχώρηση του ευρώ σε ρεαλιστικά επίπεδα και έχουμε πολύ, θετικέ επενδυτικέ επενδυτικές όπω όπως το σχέδιο juncker και την πρωτοβουλία ε, του κυρίου λαμασούρ και όσων συνεργάστηκαν μαζί του. Επομένω αλλάζει η εικόνα και διακρίνω ένα είδο αμηχανία και από την πλευρά τη αριστερά η οποία έχει την τάση να προβλέπει την καταστροφή που δεν έρχεται και από την, τάση, και από την πλευρά θα έλεγα της ακροδεξιάς των ευρωσκεπτικιστών ή των αντιευρωπαίων οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν ότι με το πέρασμα του χρόνου πηγαίνουμε καλύτερα και όχι χειρότερα. δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι αλλάζουν οι προγνώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία προς το καλύτερο δηλαδή όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και υπάρχουν χώρε μέλη οι οποίε μπορούν να δείξουν τα δικά του success stories από την πολωνία μέχρι την ιρλανδία τα οποία βέβαια δεν είναι απαλλαγμένα από οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. ευχαριστώ. Ο κύριο Φερνάντες, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι να συγχαρώ τον συνάδελφο Λαμασούρ για την εργασία του, για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι ανοίγει δρόμο για ένα νέο τρόπο ε, χρηματοδότησης για να αποκτήσουμε τις αναγκαίες επενδύσεις που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Είναι μια νέα φάση όπου θέλουμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, να μην ξεχάσουμε τα τελευταία χρόνια περικοπών, ε, προσαρμογών μια πολύ περιορισμένη αντίληψη, όπως είπε και στην Άλφος Μπερές, η οποία παρεμπόδισε την ανάκαμψη της Ευρώπης, της επενδύσεις, την απασχόληση. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτά τα ταμεία ΕΛΤΙΦ, χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια που θα συνεργαστεί ε, στα πλαίσια του σχεδίου Γιούνκερ και με το Ταμείο στρατηγικών επενδύσεων, ούτως ώστε να έχουμε επενδύσεις, ούτως ώστε το μεγάλο ποσό ρευστότητα που υπάρχει να πάει στην πραγματική οικονομία και η Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει και την ε, κεφαλαιακή ένωση, ούτως ώστε όλα αυτά τα μέσα να δημιουργήσουν ανάπτυξη στην Ευρώπη, επενδύσεις, απασχόληση πάνω απ' όλα και να ξεπεράσουμε ε, το πρόσφατο παρελθόν όπου η πλειοψηφία συντηρητική, η συντηρητική και νεοφιλελεύθερη πλειοψηφία έδρασε με τόσο απότομο και απαράδεκτο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζαμπάσκης ένα λεπτό τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα της ζωτική ανάγκης μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη για την βιώσιμη ανάπτυξη και μια ανάπτυξη που να ανταποκρίνεται στους στόχους του 2020 και να περιλαμβάνει ιδιώτες, επενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει όλα αυτά να είναι πράγματι μακροπρόθεσμα, διότι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι οι μόνες που μπορούν να αναπτύξουν την πραγματική οικονομία. Υπάρχουν και επενδύσεις βέβαια για διαφορετικού τύπου και θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του Ταμείου τα χρήματά του. Να διαχωρίσουμε τις μακροπρόθεσμες από τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. 1,5 λεπτό. Πιστεύω. Κύριε, νομίζω ότι εδώ πέρα η λέξη κλειδί είναι η συνέργεια, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Μόνο αν μπορέσουμε να επιτύχουμε την συνέργεια όλων των μηχανισμών της οικονομίας μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Και επομένως θα πρέπει να συνδυάσουμε το σχέδιο Juncker με πολιτική συνοχής, αλλά και με αυτά τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια του τώρα συζητούμε. Με τη συνέργεια λοιπόν όλων αυτών των συνιστοσών θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, αρκετούς πόρους οι οποίοι όμως θα πρέπει να διοχετευτούν στους διάβλους τους σωστούς. Πάντως θα πρέπει και οι ΜΜΕ να καλυφθούν από αυτά τα κεφάλαια. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Βιέγκας για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει να βρούμε προοπτικές ανάπτυξη. Μιλούμε για καινοτομία και σκεπτόμαστε ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν μπορούν να αποδώσουν. Εάν δεν λειτουργεί η αγορά, χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Είδατε τι γίνεται με τις τράπεζες. Γίνεται τώρα χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ύφεση θα σταματήσει με μια άλλη πολιτική. Χρειάζεται μια δημόσια επένδυση που να βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος μονό για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κράχ του 2008 ήταν ε, το αίτιο τη κρίση, που παίζει μεγάλο ρόλο ακόμη στην οικονομία. Ο κύριο Κίρτσος του ΕΛΚ θεωρεί ότι όλα πάνε καλά παρόλα αυτά. Επειδή το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δεν χρηματοδοτεί σχεδόν καθόλου τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και, τις, ε, και γενικά την πραγματική οικονομία, επειδή έχουμε όλα αυτά τα τοξικά προϊόντα, πρέπει να επανέλθουμε στη χρηματοδότηση τη παραδοσιακή οικονομία με ένα σταθερό σύστημα που, είναι, που να είναι αποσυνδεδεμένο από την κερδοσκοπία των παγκοσμίων αγορών. Το ΕΛΤΙΦ λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θετικά. Θα χρηματοδοτήσει τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όμω θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί οι κανόνε. Για παράδειγμα, το 60% για μακροπρόθεσμε επενδύσει θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκέ. Τι θα γίνει το υπόλοιπο, που υποτίθεται πω και αυτό πρέπει να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα να εξέλθει κανεί από το πρόγραμμα πριν το τέλος ε, τη χρηματοδότηση. Αυτό δεν βοηθάει τι μακροπρόθεσμε χρηματοδοτήσει. Αλλά δεν εμποδίζουμε καθόλου τους επενδυτές γήπες. Δεν υπάρχουν κανόνες. Οπότε θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και ε, γι' αυτό ακριβώς θα απόσχουμε σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ συνάλφε Μονό. Ο συνάδελφος Χέις, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κυρία Βέστα και κύριε Επίτροπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και συγχαρητήρια στον Ελένα Μασούρ για τη δουλειά του όσον αφορά αυτό το νομοθέτημα. Νομίζω ότι σε συνεργασία και αν συνδυάσουμε το Ταμείο για Στατικές επενδύσει και το πρόγραμμα Juncker θα καταφέρουμε να βγάλουμε την Ευρώπη από αυτή την τρομερή κρίση όπου έχουμε 20% των επενδύσεων που αποσύρθηκαν από το 2008 που έπεσε, που, που έπεσε έξω τέλο πάντων η Lehman Brothers. Οπότε κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό είναι να παράσχουμε μια βεβαιότητα, μια ασφάλεια στα χρηματοοικονομικά, στις ασφάλειες και έτσι να αξιστούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, γιατί αυτό θέλουν. Θέλουν βεβαιότητα ότι θα έχουν απόδοση τα χρήματά και δεν θα τα χάσουν. Και επίση βεβαιότητα όσον αφορά τις επενδύσεις που θα κάνουν. Αυτό χρειάζεται τη σήμερα ημέρα, ναι, Πρόεδρε, η Ευρώπη. Είναι απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά. Τα είπε η Επιτροπή ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να τονώσουμε τις επενδύσεις. Να πάμε κάπου μεταξύ του ενός και των δύο, τρεις ευρώ. Άρα χρειάζεται ε, να υπάρχουν αυτά τα μεδυτικά κεφάλαια, ούτως ώστε οι αγορές να ξέρουν ότι μπορούν μακροπρόθεσμα να επενδύσουν. Και, εν κατακλείδη, έχω να σας πω το ότι αν τα δημοσιονομικά εξηγένονται, τότε θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Άρα έτσι να κινούμε προς τις κεφαλαίες αγορές, γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα που μας χρειάζεται. Ευχαριστώ. Επιτρέπετε μία ερώτηση από τον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Χέιζ, επιτρέπετε να σας απευθύνει ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω. οι τράπεζες ε, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολλά προγράμματα γιατί δεν έχουν κεφάλαιο. Δεν θεωρείται ότι τα, τα προγράμματα αυτά που θα δημιουργούσαν απασχόληση και που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, δεν θεωρείται λοιπόν ότι αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το ε, πρόγραμμα Juncker. Ναι, συμφωνώ, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Juncker και αν μπορούμε να μάθουμε κάτι από τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, το χρησιμοποιούν με πολύ πιο στρατηγικό τρόπο εκεί. Γιατί τόσο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξαγοράζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνονται παγκόσμια εμβέλειας επιχειρήσεις και εμείς τις κάνουμε. Είναι λοιπόν σημαντική αυτή η χρηματοδότηση μέσω του επιχειρηματικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου υψηλού κινδύνου, venture capital. Συμφωνώ απόλυτα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίλ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, το ΕΛΤΙΦ ελπίζουμε να μπορέσει να βοηθήσει προγράμματα μακροπρόθεσμα επενδύσεων γιατί αυτό θα ήταν πραγματικά θετικό. Για μένα το σημαντικό θα ήταν να στοχεύει προγράμματα που να αυξάνουν την απασχολησιμότητα και την πραγματική οικονομία. Δυστυχώς απερίφθη το αίτημα του Κοινοβουλίου να δίνονται συστηματικά πολύ μεγαλύτερα ποσοστά χρηματοδότησης σε τέτοιες επενδύσεις. Το ΕΛΤΙΦ επίσης είναι, θα ήταν σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση των στόχων που πολλές φορές μας θέτει η Κομισιόν για την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας για να αναζωογον αναζωογονηθεί αυτή. Αλλά πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και τυποποίηση ώστε να γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές ποιοι ακριβώς είναι οι κίνδυνοι που θα αναλάβουν. Συγχαίρω την Προεδρία και τον κύριο Τραμασούρ. Διακόπτεται η ομιλήτρια γιατί τελείωσε ο χρόνος της. Λόπες Μπερμέχο. Καλημέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ακόμη να προωθήσει τη φελευθεροποίηση των κεφαλαίων ενώ έχουμε κρίση των ε, χρηματαγορών και έχουμε αυτό το νέο τύπο ταμείου επενδύσεων ένα εργαλείο που θα επιτρέπει μεγάλες ομάδες ανωνύμων επενδυτών να μπουν στο ζουμερό χώρο των δημοσίων προμηθειών. Το μόνο που μπορεί να μας, ε, να μας εγγυηθεί είναι αυτό. Οπότε θα έχουν κάθε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους όπως θέλουν. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε κάτι τέτοια, ενώ το κράτος και οι κανονικές τράπεζες θα μπορούσαν να επενδύσουν πολύ καλύτερα. Αυτή η φιλελευθερωποίηση πηγαίνει μαζί με μια ατζέντα ιδιωτικοποίησης. Εμείς δεν θέλουμε όμως οι τράπεζές μας ή τα νοσοκομεία μας να είναι στα χέρια των κερδοσκόπων. Γιατί η Ευρώπη δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι στα χέρια αυτών αλλά των εργαζομένων. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Ενάμιση λεπτό ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών Είμαστε διατεθειμένοι στον τομέα των υποχρεώσεων να δείξουμε ευελιξία, αλλά όχι στον τομέα των πληρωμών. Μπορού, πολλά μπορούμε να κάνουμε με το front loading για να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση, αλλά όταν θα φτάσουμε στην αναθεώρηση θα πρέπει να δούμε από πού θα έχουμε φρέσκο χρήμα για να εφαρμόσουμε αυτά που προβάλλονται. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη να δίνουν άδειες διασυνοριακές. Για παράδειγμα, για τις ε, συχνότητες κινητής τηλεφωνίας. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι προκηρύξεις και οι διαγωνισμοί να γίνονται την ίδια μέρα και τα ποσά που θα έχουμε έτσι να αξιοποιούνται για να κάνει επενδύσεις, ε, να το έχουν ως κεφάλαιο για επενδύσεις τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά όργανα ε, για να χρηματοδοτούν προγράμματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ή για να μειωθούν οι εκκρεμούσες πληρωμές ούτως ώστε να τις αξιοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις για να αναπτύξουμε τις υποδομές μας και να επιτρέψουμε στο μέλλον να γίνουν ακόμη περισσότερες πληρωμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. 1,5 λεπτό ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμασούρ, η έκθεσή σας αξίζει της υποστήριξής μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Αναφέραμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μια που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ενιαία αγορά και εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ας μην στρέφουμε την προσοχή μας στις διαφορές μας, αλλά σε αυτά που μπορούμε να συνεργαστούμε. Μπορούμε να λιάνουμε αυτές τις διαφορές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την κοινοτική μέθοδο. Άρα, να προχωρήσουμε σε αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για μένα. Και είμαστε υπέρ της πραγματικής οικονομίας και των επενδύσεων μέσα στην επενδυτική οικονομία, ακριβώ όπω τα είπε ο κύριο Ρούμπιχ. Επενδύσει χρειάζονται στι υποδομέ και στι μεταφορέ δηλαδή. Οπότε μπορούμε να φτάσουμε στα 400-500 δις με το 2020. Έχουμε προϋπολογισμό 36 δι. Οπότε έτσι μπορούμε να γυφρώσουμε τις διαφορές μας χρησιμοποιώντας τα ομόλογα έργων. Αυτό θα ήταν μια άριστη λύση. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Η κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμασούρ για την εξαιρετική του εργασία επί του ΕΛΤΙΦ που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξη και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύω όμως ότι αυτό το επενδυτικό ταμείο είναι κάτι που θα έπρεπε να συμπληρώνει τη χρηματοδότηση, την παραδοσιακή χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να επεξεργαστούμε τις ε, κανόνες που θα ισχύουν για τη λειτουργία των τραπεζών. Έχουν επιβληθεί ορισμένοι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το τραπεζικό σύστημα θα λειτουργεί υγιώς και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων που χορηγείται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή. Το 70% των ετοιμάτων για δανεισμό χορηγείται με επιτόκιο περίπου 2,7% άρα το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί λίγο πολύ σωστά αλλά παρόλα αυτά στην Ευρώπη γινόμαστε όλο και περισσότερο ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις διότι υπάρχουν επενδυτές που ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Βίρκουνεν, Ενάμιση λεπτό. Ο Ζάλφος Ουγέλβη. Πρόεδρε, δεν είμαι ευρωσκεπτικιστής. Δεν θέλω να γκρεμίσουμε την Ευρώπη μας. Είμαι μέλος των σοσιαλδημοκρατών και πιστεύω σε μια ενωμένη Ευρώπη. Δεν θα πρέπει όμως να εθελοτυφλούμε. Θα πρέπει να βλέπουμε κατά πρόσωπα τα προβλήματα. Γι' αυτό και θέλουμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη χωρίς μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Μιλούμε για 5,5 εκατομμύρια νέους ανέργους. Μιλούμε για νέους της γενιάς μου. Κατά εκατοντάδες χιλιάδων φεύγουν από τη χώρα, γιατί στην Ουγγαρία δεν βρίσκουν δουλειά. Θα πρέπει η Ενωμένη Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει να αναζωογονήσουμε τη βιομηχανία της Ευρώπης και να μην γίνουμε ουραγοί. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι βοηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επομένω, να έχουμε μια ισχυρή οικονομία που να δημιουργήσει απασχόληση, μια ασφαλή κοινωνία. Εγώ σας υποστηρίζω. Θα πρέπει επομένω οι πόροι αυτών των κεφαλαίων να χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη, αλλά όχι για κερδοσκοπία. Και να μην ξεχνάτε την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Να μην έχουμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων Οπότε ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχει αυτή η πρόταση. Κύριε Ουελή, δέχεστε μία ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Κόψιτς. Αγαπητέ συνάδελφε, μιλήσατε για την αργία των νέων και την ανάγκη επαναβιομηχάνησης της Ευρώπης. Δεν θα συμφωνούσατε ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς όπου χρειαζόμεθα μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το έχουμε ήδη συζητήσει. Και θα ήθελα οι συναδέλφοι να με ακούσουν. Γιατί δεν ασχολούμεθα επαρκώς με τον τουρισμό που συνδέεται με την ανεργία των νέων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ καλή ερώτηση από τον ε, Κροάτη συνάδελφο Ευχαριστώ πολύ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός χρειάζεται μακροπρόθεσμες επενδύσεις μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες και μακροπρόθεσμα και μπορεί να δώσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και υπάρχει, όπως ξέρετε, παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον τουρισμό και η Ευρώπη ε, βραδιπορεί, γιατί δεν έχουν γίνει επαρκείς επενδύσεις. Και αυτό είναι επίκριση και για το πρόγραμμα Juncker, γιατί δεν περιλαμβάνεται ο τουρισμός ε, στον, ε, στους στόχους του. Ο η συνάδελφος Νταντσίλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε έναν όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε όλο ένα και περισσότερο χρήμα που θα μπαίνει στην πραγματική οικονομία και τις ροές στην αγορά. Οπότε Έχουμε τώρα κάποια ρευστότητα, αλλά δεν είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά τι μακροπρόθεσμε επενδύσει, γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη εμπιστοσύνη από του επενδυτέ. Άρα η πρόκληση είναι το πώ θα μπορέσουμε να γίνουμε ελκυστικοί για τι ιδιωτικέ επενδύσει. Είναι κάτι που το χρειάζεται η Ευρώπη. Πρέπει να ρισκάρουμε για να ελκύσουμε του επενδυτέ να προβούν σε μακροπρόθεσμε επενδύσει. Όπω στι τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, τι μεταφορέ, στην παιδεία, και όλα αυτά να γίνουν μετοχές, τοκομερίδια κλπ. Οπότε έτσι θα γίνει η Ευρώπη και έτσι θα έχουμε θέσει απασχόληση Θεωρώ θετική την πρόταση της ε, Επιτροπής για το να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. δεν υπάρχουν εσωτερικέ συνόρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι ιδιώδη αγορά. Και αυτό θα ωφελήσει και τι παραμεθόρε περιοχέ τη Ευρώπη και όλου. Η συνάδελφο Καηλή, 1,5 λεπτό. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων και εκφράζω την πεποίθησή μου ότι αυτό το όχημα επενδύσεων για εναλλακτικέ επενδύσει είναι το κατάλληλο για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ευρώπης σε περιουσιακά στοιχεία ανάπτυξης αντίθετα από το πρόγραμμα Juncker που είναι αντικυκλικό και δεν λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της απομόχλευσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορεί να επιτύχει υψηλότερο πολλαπλασιαστή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση για να ασχοληθεί περισσότερο με την ε, προσφορά μεταξύ των περισσιακών στοιχείων που θέλει να επενδύσει εδώ πρέπει να είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις δυνατότητες επενδύσεων και να ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς θα αποδοθεί το χαρτοφυλάκιο αυτών των επενδύσεων και να στοχεύσουμε όχι μόνο στις μικρομεσαίες αλλά και σε γεωγραφική κατανομή χωρίς βέβαια να στρεβλώνουμε τις επενδύσεις και λαμβάνοντας υπόψη και τις νομικές δομές του Ευρωπαϊκού Νότου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Καϊλίν. Ένα λεπτό. Η κυρία, ο κύριος Μπαγιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Λαμασούρ για την έκθεση του. Αυτό το Ταμείο Μικροπρόθεων Επενδύσεων θα είναι ίσως ένα κατάλληλο πλαίσιο για να επιτρέψει στις επενδύσεις σε πραγματική οικονομία αν και θα ήθελα να θυμίσω ότι εμείς δίνουμε σημασία ε, η σοσιαλιστική ομάδα και σε πολιτική επενδύσεων αποπληθωριστικών, ε, κατά του αποπληθωρισμού μάλλον. Να επανέλθω στο ΕΛΤΙΦ λοιπόν. Θα ήθελα να θέσω ορισμένες κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν οι κερδοσκόποι που εκμεταλλεύονται την κεφαλαία αγορά. Επίσης χρειάζεται σαφέστερος ορισμός για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για υποδομές στο θέμα των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Εννοούμε παραγωγικές υποδομές και όχι μη παραγωγικές όπως ας πούμε τα, τις αγορές κτηρίων από ταμεία που δεν είναι παραγωγικές. Επίσης η τοποθέτηση των ε, επενδύσεων πρέπει να μην είναι στους φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στάλφεν. Δεν βλέπω τον κύριο Γκουαλτιέρη. Οπότε πρέπει στη διαδικασία προσέλκυση. Ε, α, συγγνώμη, πριν τη διαδικασία προσέλκυση προσοχή του Πρόεδρου, θέλω να πω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων χθε το βράδυ ενέκρινε μια έκθεση για την άρση της ασυλίας του κυλίου Στάνη.